είναι μια διαδικασία, μια διεργασία και όχι ένα συμβάν μεμονωμένο. εισαγωγή του ευρώ. Έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας, έχουμε τη συνθήκη ε, για τις δημοσιονομικές ισορροπίες, το μηχανισμό σταθερότητας, ε, το μηχανισμό για την καταπολέμηση οικονομικών ισορροπιών, τη συνθήκη για το ευρώ. Βέβαια παραμένουν, όπως είπατε και εσείς, πολλά να γίνουν. Το ε, γνωρίζει πολύ καλά και ο Μάριο. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε ε, την οικονομική, τη χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση και εγώ, αν μου επιτρέπετε ένα προσωπικό σχόλιο, θα πρέπει να δοθεί σάρκα και οστά ε, στον προϋπολογισμό, να γίνει σημαντική πρόταση με την ε, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, να υπάρξει ένας υπουργό Οικονομικών στην Ευρωζώνη και τέλος να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση της ΩΝΕ. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα για να δοθεί ο τελευταίος λόγος προς αυτό και στους ευρωβουλευτές φυσικά. Βέβαια, μιλώ για τους βουλευτές ε, που εκπροσωπούν ε, τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Καταθέτω ότι και στις ακροάσεις που είχα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα την πιο ένθερμη ηθική υποστήριξη ε, για τη σταθερότητα αλλά και για μέτρα γενναία τολμηρά μη συμβατικά όπως αγορά ε, περισσοκών στοιχείων κάποιων το 2010-2011 πριν ληφθεί απόφαση από την ΕΚΤΑ υπό τον Ντράγκη για, τη, για τα επόμενα μέτρα πρέπει ε, να είστε πιστοί στην εντολή σας και να δίνετε ε, σταθερότητα ε, στις τιμές, να είστε τολμηροί όταν πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις σας και να έρεστε στο ύψος των ευθυνών σας. Αυτή ήταν η εντολή που μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέποντας το Ευρωβαρόμετρο, και βλέποντας την εμπιστοσύνη ε, που δείχνουν οι πολίτες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα ξεπερνά ε, την έλλειψη εμπιστοσύνης και είναι καλύτερο το αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε για τα Εθνικά Κοινοβούλια και το λέω εμπαρόδο και με πολύ προσοχή. Κανείς δεν μπορεί να πει ε, σήμερα ε, ποια θα είναι η μορφή ε, της αλλαγής ε, γιατί αλλάζει το μέλλον με τις προκλήσεις που είναι σήμερα απρόβλεπτες. Αυτό είπε ο Ζαμονέ και παραμένει επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Πρέπει να σας πω μας κύριε Πρόεδρε ότι αυτό που ήδη ξέρουμε είναι ότι η Ευρώπη το αύριο θα υποφεληθεί από αυτό το αξιόπιστο νέο νόμισμα που έχει από το ευρώ δηλαδή αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ε, την χάνει τη πλούσια εμπιστοσύνη των πολιτών. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Και τώρα το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Μάριο Ντράγκη. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, αγαπητέ Jean-Claude, ε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Ε, με μεγάλη ικανοποίηση βρίσκομαι εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε από κοινού την πρώτη 20 του ευρώ. Ε, το ευρώ είναι η πιο απτή εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ε, είναι το το σύμβολο που χρησιμοποιούν καθημερινά οι Ευρωπαίοι πολίτε αυτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και είναι σημαντικό που, και κατάλληλο που εορτάζουμε εδώ αυτή την 20η επέτειο του ευρώ με τους άμεσα ερετούς εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών. Και μάλιστα εδώ οι άμεσα αιρετοί εκπρόσωποι και οι ηγέτες ε, και οι αιρετοί εκπρόσωποι και σε άλλα κοινοβούλια πολύ σωστά αναγνώρισαν ότι η εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας και της οικονομικής σταθερότητας μακροπρόθεσμα είναι μια κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζεται συλλογικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί εν τη Με την ενία αγορά έχουμε ένα ισχυρό μηχανισμό βιώσιμης ανάπτυξης για να στηρίξει το βιωτικό μας επίπεδο και τις βιωτικές μας συνθήκες. Η Ευρώπη διαφύλαξε την ακεραιότητα της ενίας αγοράς και το ευρώ το ίδιο. Σήμερα η οι οικονομίες μας ε, είναι ολοκληρωμένος ε, σε βαθμό αδιανόητο όταν πρωτοσχεδιάστηκε το ευρώ. Οι ενδοευρωπαϊκές ε, εξαγωγές πέρασαν το 15% στο 20% του ΑΕΠ σήμερα αλλά κυρίως οι αλυσίδες αξιών παντού σήμερα στην Ευρωζώνη ε, είναι υψηλότερες. Το ευρώ μάλιστα είχε και δύο δεκαετίες ε, σταθερότητας τιμών, ακόμη και σε χώρες που κάτι τέτοιο ήταν ε, παλιά ανάμνηση. Σταθερές τιμές ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη του κόσμου στην αξία των αποταμιεύσεων του των οικονομιών του, Κάτι που είναι προϋπόθεση για την ευημερία. Και με βάση αυτή την εμπιστοσύνη, οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν επενδύσει και να δημιουργούν θέσεις απασχόληση. Σήμερα οι περισσότερες προκλήσεις έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά. Και αυτή η συνεργασία, αυτή η συλλογικότητα μεγενθύνει την ικανότητα των μεμονωμένων χωρών να διασφαλίσουν την εθνική τους κυριαρχία στα σημαντικά ζητήματα. Γιατί αυτή η εθνική κυριαρχία διαφορετικά θα είχε διαλυθεί, θα είχε χαθεί μέσα στο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Και ακριβώς γι' αυτό το ενιαίο νόμισμα έχει δώσει σε όλα τα μέλη της Ευρωζώνης την κυριαρχία στις νομισματικές τους πολιτικές σε σχέση με τις προϋπάρχουσες νομισματικές ρυθμίσεις. Και από κοινού έχουμε καταφέρει να έχουμε στεντόρια φωνή και σημαντική φωνή στη ρύθμιση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών. Μία φωνή μάλιστα που είχε κέριο ρόλο στη διαμόρφωση της, ε, των ρυθμίσεων των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών μετά την ε, χρηματοπιστωτική κρίση, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Βέβαια, σε κάποιες χώρες δεν έχουν υλοποιηθεί στο έπακρο όλα τα πλεονεκτήματα του ευρώ. Και εν μέρει οφείλεται αυτό στο ότι οι μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητες και κάτι τέτοιο θα ίσχυε σε οποιοδήποτε νομισματικό σύστημα. Τέτοιε μεταρρυθμίσει είναι απαραίτητε για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Εν μέρει επειδή η Οικονομική και Νομισματική ε, Ένωση εξακολουθεί να είναι ατελής ή ημιτελής. Σημαντική πρόοδος βέβαια έχει συντελεστεί από την έναρξη της κρίσης, αλλά θα πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας και δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Στο μέλλον όλοι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για να καταστήσουμε την Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση μια, έναν ακόμη ισχυρότερο μηχανισμό ευημερία για όλα τα κράτη-μέλη της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε, έχει και θα έχει θεμελιώδη ρόλο στην καθοδήγηση και στο σχεδιασμό του ευρωπαϊκού μας μέλλοντος. Και στο παρελθόν, από κοινού με τους Ευρωπαίους ηγέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε θεμελιώδεις αποφάσεις για την δημιουργία της ενιαίας αγοράς και για την δημιουργία και την ε, ίδρυση του ευρώ. Και σήμερα όλοι δρέπουμε τους καρπούς αυτής της δέσμευσης, της δέσμευσης και της στράτευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτό το στόχο. Και θέλουμε και οι μελλοντικέ γενναίε των Ευρωπαίων να υποφεληθούν από τη δική μα δέσμευση και τη δική μα στράτευση στα θέματα αυτά. Σήμερα, καθήκον μα είναι να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε πριν από δύο δεκαετίε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα να δώσω αμέσως το λόγο στον Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζαν Κλοντ Juncker. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση έκπληξη. Πρέπει να θυμηθείτε ότι κάποιοι από εσά όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία προς το ενίο νόμισμα μας θεωρούσατε ότι είμαστε τρελοί και λέγατε ότι επουδενή αυτή η νομισματική ένωση μεταξύ τόσων διαφορετικών χωρών δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Τους ακούμε λιγότερο σήμερα αυτούς. Κάποιοι βουλευτές εδώ και εκεί, δημοσιογράφοι, παρτού, παντού, ε, νομικοί, καθηγητές δικαίου κυρίως στη Γερμανία, οικονομολόγοι στη Γερμανία, όλος ο κόσμος έλεγε ότι κινούμεθα προς μια περιπέτεια που θα οδηγούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο χείλο της Αβίσου. Πόρα απέχουμε από την Άβυσο, διότι σήμερα διαπιστώνουμε με θικανοποίησο και σχεδόν με ευτυχία ότι το έργο που αναλάβαμε και ξεκινήσαμε εδώ και 20 χρόνια εστέφθη από επιτυχία. ήταν εκτελικά νίκησαν αυτοί που έβλεπαν προς το μέλλον, όπως δύο προκάτοχοί μου. Ο Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, ο Πιέρ Βέρνερ, ήταν από αυτούς. Χωρίς τη φαντασία εκείνου του ανθρώπου τίποτα δεν θα ήταν δυνατόν. Και με αναφέρω και τον Ζακ Ντελόρ, που ήταν ε, υπέρμαχος της ευρωπαϊκής οικονομικής αυτής ε, προσπάθειας. Θα μπορούσα να προσθέσω και άλλα ονόματα σε αυτά, πολύ άριθμα. Αλλά όχι τόσα πολλά ονόματα όσο εκείνοι που πίστευαν ότι πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι πρέπει να γίνει αυτό το εγχείρημα. Εγώ ήμουν υπέρ της περιπέτειας που εστέφθη τελικά από επιτυχία μαζί με άλλους, με τον Jean-Claude Trichet, σαν πρόεδρος της διακυβερνητικής διασκέψεως το 1991, ηγηθήκαμε της διαδικασίας που μας οδήγησε στη συνθήκη του Μάστριχτ. Το τμήμα το νομισματικό του Μάστριχτ είναι ένα πετυχημένο τμήμα, ενώ το πολιτικό τμήμα της συμφωνίας του Μάστριχτ ήταν πιο αδύναμο, θα έλεγα μέτριο. Και θεωρούσα τότε όταν υπέγραφα τη συνθήκη του Μάστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου του 1992 και ήμουν ο μόνος που είχε απογράψει τη συνθήκη που και που ζει ακόμα, είναι ζωντανό στην πολιτική ζωή. Ε, πίστευα τότε ότι η λογική και ο δυναμισμός του ενιαίου νομίσματος θα μας οδηγούσε προς εμβάθυνση της πολιτικής ένωσης. Μεγάλη ε, απογοήτευση, διότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Όπως και η σύγκληση, η οικονομική και κοινωνική, μεταξύ διαφόρων κρατών μελών, της ε, Ευρωζώνης. Αυτή ε, δεν έχει επιτευχθεί όπως τα θέλαμε. Πάντα θεωρούσα ότι βασικό πλεονέκτημα της το βασική, βασική συνιστός επιτυχίας του νήμου Μήμπορτος ήταν από την ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν τον Ιανουάριο του 1991 και θέλαμε αυτή την ανεξαρτησία από τότε διότι αυτό δίνει αξιοπιστία στο ενίο νόμισμα. Δεν αμφισβητήθηκε αυτό ποτέ η αξιοπιστία του νομίσματος ούτε από τις αγορές. Κάποιος να παίρνει τηλέφωνο, δεν ξέρω, κάποιος Γάλλος. Α, τώρα ξέρω. Η μεγάλη συζήτηση, το βασικό θέμα ρίχνει τη σκιά του παντού. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα ήταν ανεξάρτητη, δεν θα τα πετυχαίναμε αυτό. Εμεί πολεμήσαμε για την ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χωρί αυτή την εξαρτησία δεν θα ήταν επιτυχία το νέο νομισμα, την επιτυχία που έχει σήμερα. Υπάρχουν και δυναμίε βέβαια. Εγώ ανήκα σε εκείνου μαζί με τον Τελόρ και τον Μέστατ και τον Μπερεγκοβουά που από την αρχή θέλαμε να υπάρχει οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Είναι μια μεγάλη αδυναμία αυτή για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, που δεν είναι τέλειος ο συντονισμός. Ποτέ δεν ήταν τέλειος συντονισμός. Έπρεπε να κάνουμε όμως περισσότερο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και δημοσιονομικών και φορολογικών. Αυτή η δυναμία παραμένει και δεν μπορούμε να παρετηθούμε, αλλά θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να τα προσεγγίσουμε αυτά, να τα συζητήσουμε που είναι πολύ σημαντικά για το εγχείρημα που έχουμε μπροστά μας, για την οικοδόμηση που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί επέκριναν την πολιτική της Ευρωζώνης. Το παίρνω αυτό προσωπικά, διότι ήμουν πρόεδρος του Eurogroup όταν μας έπληξε μεγαλύτερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Πράγματι, επευλήθη ε, λιτότητα με τρόπο κάπως απρόσδεκτο. Δεν είχαμε αναλύσει πολύ ε, την πολιτική. Όχι γιατί θέλαμε να τιμωρήσουμε εκείνους που ήταν στην ανεργία και που εργαζόταν, αλλά διότι οι διαθροτικέ μεταρρυθμίσει, ανεξάρτητα από τον νομισματικό καθεστώ στο οποίο βρίσκεται κανεί, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικέ. Λυπούμε, διότι δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία στην επιρροή που είχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πολύ όταν ξέσπασε η κρίση, πιστεύαμε ότι η Ευρώπη είχε επαρκείς δυνάμεις για να μπορεί να αντισταθεί μόνη της χωρίς την επιρροή του Δούνου του και να αντιμετωπίσει αυτή την ε, κρίση. Αν η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει δυσκολίες, οι ΗΠΑ δεν στρέφονται προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά προς τις ΗΠΑ Πολιτείες της Αμερικής. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε κι εμείς. Επίσης, πάντα με έθλιβε αυτή η έλλειψη αλληλεγγύης που διαπιστώθη όταν ξέσπασε η ελληνική κρίση, όπως την αποκαλέσαμε δεν ήμασταν ε, επαρκώς αλληλέγγυοι έναντι της Ελλάδας. Και χαίρομαι διότι βλέπω ότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία και άλλες χώρες έχουν ξαναβρει. Δεν θα έλεγα μια θέση στον ήλιο, αλλά μια θέση ανάμεσα στις ε, υγιείς ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Και δεν μπορώ να τα πω όλα ε, τώρα, ε, γιατί θέλω να σας αφήσω λίγο να περιμένετε τα απομνημονεύματά μου ε, και εκεί θα πω τα υπόλοιπα. Αλλά παραμένω της άποψης πως η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση ουσιαστικά είναι μια πολιτική υπέρ της ελευθερίας Και γι' αυτό, στο όνομα της δικής μου γενιάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ε, κατέστησαν ε, δυνατή την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και το ευρώ που είναι η μόνη συμβολή, θα έλεγα το μόνο λιθαράκι ε, της ε, δικής μου γενιάς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν πολλά λάθη. Εμείς είμαστε παιδιά που γεννηθήκαμε από τον πόλεμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χέλμουτ Κόλ. Χωρίς αυτό δεν θα είχε γίνει τίποτε από όσα έχουμε καταφέρει ως γενιά. Ο Χέλμουτ Κόλ και ο Τέο Βάγγελ χρειάστηκε να επιβάλλουν, να πείσουν τους Γερμανούς ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, για το ευρώ. Το ίδιο ε, χρειάστηκε να κάνουν και άλλοι. Ο Βιμ Κόκ, για παράδειγμα, που επίσης πρόσφατα πεβίωσε άλλωστε, επίσης έκανε πάρα πολλά και πρέπει να μείνουμε πιστοί στη μνήμη τους και στο έργο τους. Merci ευχαριστώ πολύ, Jean-Claude. Και τώρα θα ακούσουμε τη δήλωση του κ. Σεντένου, Προέδρου της Ευρωομάδας. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε της ευρωπαικης Κεντρική Κεντρικής Τράπεζας, αγαπητέ Jean-Claude Trichet, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Με ιδιαίτερη χαρά γιορτάζω μαζί σας την 20η επέτειο από την εισαγωγή του ευρώ. Το ευρώ είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το νέο μας νόμισμα είναι μια σταθερή άγκυρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για την ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το ευρώ είναι σύμβολο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. σε 19 χώρες Ευρωζώνης 340.000 ε, πολίτες ε, το χρησιμοποιούν και το υποστηρίζουν. Είναι το δεύτερο πλέον χρησιμοποιούμενο νόμισμα και έτσι ενισχύει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο προσκήνιο. Πολλοί προέβλεπαν ε, μια παταγώδη αποτυχία του ευρώ, όμως αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Τα τελευταία 20 χρόνια πράγματι δεν ήταν εύκολα στο σύνολό τους. Είχαμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, τη κρίση του δημοσίου χρέους ε, που δοκίμασε το ευρώ. Υπήρξαν ελλείψεις και αδυναμίες ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, που ανέκυψαν. Ωστόσο, βγήκε πιο ισχυρό το νόμισμα του ευρώ από την κρίση και δεσμεύτηκαν οι πολιτικοί για την ανάληψη δράσης και για την τροποποίηση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα, Τραπεζική Ένωση που ενισχύουν και τον οικονομικό συντονισμό και δείχνουν ακριβώς αυτή τη βούληση των πολιτικών. Η Ευρωζώνη σήμερα βρίσκεται σε επεκτατική φάση. Αυτό ξεκίνησε το 2013. Έχουμε θετικές προοπτικές και εκτιμήσεις παρά τους κινδύνους ε, και ορισμένοι από τους συσσωρεύονται. Βλέπουμε αύξηση των θέσεων εργασίας, άρα όλο και περισσότεροι ωφελούνται από την επέκταση, από τη μεγέθυνση. Τα δημόσια οικονομικά, ο τραπεζικός τομέας επίσης ε, σημειώνουν βελτίωση. Πολλά επίσης ε, στους στα 27 χρόνια, αλλά και πολλά πρέπει να γίνουν ώστε να εξοπλιστεί επαρκώς ε, η ΟΝΕ και να μπορεί να αντισταθεί σε μελλοντικέ κρίσεις. Το Δεκέμβριο στην ε, Σύνοδο Κορυφή ελήφθη σημαντική απόφαση για την ενίσχυση του ενιαίου νομίσματος με τη μεγαλύτερη δυνατή μεταρρύθμιση του ευρώ εκτός ε, πλαισίου κρίσης. Πρόκειται για μια συμφωνία που θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη ευρύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και το σύστημα ε, της ε, εγκαθάριση τραπεζών θα είναι πιο αξιόπιστο. Οι ηγέτες επίσης αποφάσισαν να, να υπάρξει και ένα δημοσιονομικό εργαλείο για τη σύγκριση και, σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι αυτό το project θα κάνει πιο σταθερή την Ένωση, μια Ένωση για όλους. Προτεραιότητά μας στους επόμενους μήνες είναι να επεξεργαστούμε αυτό το φάκελο, θα συνεχίσουμε όμως να εργαζόμαστε και ε, πάνω σε άλλα σημαντικά ζητήματα όπω είναι το σύστημα καταθέσεων η ρευστότητα και η ε, καθάριση. Βήμα-βήμα μεγαλώνουμε την ανθεκτικότητα, βελτιώνουμε την ομαλή λειτουργία ε, της ε, Νομισματικής Ένωση. Έτσι, οι χώρε τη Ευρωζώνη, οι πολίτε των χωρών τη Ευρωζώνη θα είναι σε καλύτερη θέση να δρέψουν του καρπούς του ενιαίου νομίσματο και τα επόμενα 20 χρόνια, αλλά και περισσότερα. Δεν κουράζομαι παραλαμβάνω ότι η Ένωση ε, ποτέ δεν ήταν αυτός σκοπός, ούτε το ευρώ είναι ένας αυτός σκοπός, ποτέ δεν ήταν, είναι ένα εργαλείο για μεγαλύτερη ευημερία των λαών της Ευρώπης και δική μας ευθύνη είναι να ε, τηρηθούν οι υποσχέσεις ε, ιδίω αυτούς τους αβέβαιους καιρούς. Δικό μας χρέος, δικό μας καθήκον είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία πιο ευημερούσα, πιο αλληλέγγυα, μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες εντός αλλά και μεταξύ των κρατών μελών που την απαρτίζουν. Και σήμερα ε, θα σταματήσω ε, με μια επιθυμία μου ε, να ζήσει το ευρώ, μια ισχυρή Ευρώπη. Ζήτω ισχυρή Ευρώπη, ζήτω το ευρώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα κλείνοντας τελευταία παρέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού, του κυρίου Γκουαλτιέρη. Αγαπητοί Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της Επιτροπής ΕΚΟΝ θα ήθελα να αποτίσω πρώτα απ' όλα φόρο τιμής τα πρώην κοινή μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέβαλαν στην επιτυχία του ευρώ και στην ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και της δημοκρατικής του νομιμοποίησης. Θα ήθελα ιδιαίτερως ε, να δώσω τα εύσχημα στους προκατόχους μου, τον Καρφον Φόγκαου, την Κρίστα Ράτσιο Πλάκ, την Περβάς Πέρες, τη Σάρον Μπόλς και χαίρομαι που οι περισσότεροι είναι παρόντες εδώ σήμερα και παρούσες. Από το σχεδιασμό του, το ευρώ ήταν ένα ισχυρό οικονομικό εργαλείο και ένα φιλόδοξο πολιτικό σχέδιο. Καταρχήν, το ενιαίο νόμισμα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της ενιαίας αγοράς. Ε, και χάρη στο ενιαίο νόμισμα ε, έγινε δυνατή η εμβάθυνση της ε, ενιαίας αγοράς και η ενίσχυση των οικονομιών και των αλυσίδων αξιών. Δεύτερον, όπως είπε ο κύριος Δράγκη, το ευρώ είναι προϋπόθεση για τη διαφύλαξη και την ανάκτηση της κοινή νομισματικής κυριαρχίας μετά την κρίση της τάξης του Μπρετον και την ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερως για τις πλέον ευάλωτες χώρες μέλη. Τρίτον, το ευρώ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας ειρηνικής και στενότερης Ευρώπης και Ευρώπη που θα είναι παγκόσμιο παράγοντας μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και της Γερμανικής Επανένωση. Και ουδέποτε δεν πρόκειται να ξεχάσουμε το όραμα και το θάρρος του Χέλμουντ Κόλ, του Φρασά Μιτεράν και του Ζακ Ντελόρ. Με άλλα λόγια, ένα ισχυρό ευρώ αποτελεί εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση για την προστασία, την υπεράσπιση και την ε, ε, όθηση, την επαναπρόθεση του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου, που θα πρέπει να αντιμετωπίζει ε, τι ρηξικέλευτε μεταρρυθμίσει των καιρών. Και πριν από 20 χρόνια, όταν εορτάζαμε το ευρώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η χρηματοπιστωτική κρίση θα έσυε τα θεμέλια του. Η κρίση αυτή μας ε, έδωσε δύο μαθήματα. Το πρώτο είναι ότι παρά την τέλειά της, το σθένος και η αθεκτικότητα του ευρώ ε, έχουν τις ρίζες του στην κοινή ε, πολιτική αποφασιστικότητα να διαφυλαχθεί η ακαιρεότητά του. Επίσης, ο ρόλος του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Προέδρου της είχαν αποφασιστική σημασία και το ευρώ προστάτευσε τους ευρωπαϊκούς λαούς στη διάρκεια της Κρήτης. Και Επίση, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ του ευρώ και των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια τη κρίσης, ακόμη και κάποιων λαθών οικονομικών πολιτικών που διαπράχθησαν την εποχή της κρίσης. Το δεύτερο δίδαγμα είναι ότι αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξου στόχους μας, δεν αρκεί η ανθεκτικότητα. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε το κοινό μα νόμισμα με, ε, ένα, με μια στεναρή δημοκρατική, οικονομική και κοινωνική ένωση. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε μια νέα κρίση για να αναπτύξουμε τα απαραίτητα εφόδια ώστε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ε, ευημερία όλων των πολιτών μας. Η Ευρώπη είναι ένα ταξίδι και ήρθε ο καιρό να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και είμαι βέβαιος ότι και αυτό και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκπληρώσουν στο έπακρο το καθήκον τους. Και τώρα από το κουαρτέτο Αβένα θα ακουστεί ο ευρωπαϊκός ύμνος.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 Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στις ψηφοφορίες. Απλώς να σας επισημάνω ότι έχουμε σημειώσει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, οπότε αν ζητάτε το λόγο μόνο για διαδικαστικά βάσει του εσωτερικού κανονισμού. Και ακόμη και αυτά παρακαλώ είναι πολύ σύντομα. Ο κύριος Γκόρνη έχει το λόγο. Να υπενθυμίσω κάτι στην Ολομέλεια. Ένας πρώην συνάδελφος ο πρώην Ευρωβουλευτή Έντζο Ερμίνιο Μπόζο που χάθηκε, ένα γεννόδο άνθρωπο, πρώην αστυνομικό, που είχε αφιερώσει την πολιτική του μάχη στην προάσπιση των ανθρώπων των βουνών. Να, τον θυμηθούμε και θέλω να πω αγαπητέ Ερμίνιο, εσύ πέθανε αλλά δεν πεθαίνουν οι ιδέε σου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μποργκέτσιο ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Άρθρο 25 και άλλα άρθρα του εσωτερικού κανονισμού για την εφαρμογή του καταστατικού. Το 1974, για παράδειγμα. Στις 10 Δεκεμβρίου το Προεδρείο αποφάσισε και πάλι να παρατείνει μέχρι τα 65 το θέμα της επικουρικής άδειας και να μειώσει κατά 5% το ύψος αυτής της επικουρικής άδειας χωρί τη αριθμική αναπροσαρμογή και μάλιστα ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα ακόμη πιο φιλόδοξε προσπάθειε. Βέβαια, είναι πανίσχυρος ο Γενικό Γραμματέα και η δική του ε, η σύνταξη βρίσκεται στο απειρόβλητο. Να μην σας, ε, ε, να σας υπενθυμίσω ότι το 1990 δημιουργήθηκε αυτή η επικουρική σύνταξη και για 10 χρόνια καταβάλαμε πολύ σημαντικές εισφορές και μάλιστα με προοπτικές που αναφερόνται στα επίσημα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ήδη είχαν φυγεί τα κεκτήμενα δικαιώματα το Μάρτιο του 2009, αλλά τότε μας είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα άλλαζε τίποτα περαιτέρω. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν οικονομικέ δυσκολίε σε αυτό το συνταξιδοτικό ταμείο, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φταίει. Γιατί όταν ε, υιοθετήθηκε το νέο καταστατικό των Ευρωβουλευτών το 2009, αποφασίστηκε να μην δίνονται εισφορέ στο συνταξιδοτικό ταμείο. Η λογική ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει το καθεστώ αυτό που το δημιούργησε μόνο του. Πολλά δε μάλλον που σήμερα η, ε, ευρωβουλευτές που επωφελούνται από το νέο καθεστώς δεν έχουν καταθέσει ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα ευρώ ε, ε, εισφοράς για πάρα πολλά χρόνια. Ε, μέχρι πού θα πάει η παραβίαση των κεκτημένων δικαιωμάτων των ευρωβουλευτών, πώς είναι δυνατόν να θέλουμε να υποστηρίξουμε την υπόλοιψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θίγοντας τα δικαιώματα των πιο παλιών ευρωβουλευτών. κάτι δεν θα το δεχόταν ο, οι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα που επισημάνατε. Ε, πάντως το σημειώνω και θα λάβετε απάντηση. Κύριε Άντερσον. Πρόεδρε, σύμφωνα τον ιστορικό κανονισμό άρθρο 2245 θέλω να ευαισθητοποιήσω τους ακούγοντες ε, για έναν εξάχρο, τη Λέιλα Γκέρβιν, έξι, χρόνια βουλευτήνα, που είναι σε απεργία σε 69 ημέρες, συνελήφθη πριν από ένα χρόνο διότι καταδίκασε την εισβολή της Τουρκίας στα Αφρίν. Πολλοί ευρωβουλευτές εδώ επίσης το καταδίκασαν αυτό, αλλά σε απεργία πείνας κατά της απομόνωσης των μιας γυναίκας των Κούρδων. Και κοιτάξτε την η δίκη της για την απομόνωση του Τσαλάν. Και είναι σε απεργία πείνας. Ε, ε, υπάρχει διακοπή, διακόπτει ο Πρόεδρος η κυρία Μπιλμπάου. Και αυτή είναι η τελευταία ομιλία για διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω κατάχρηση της γενναιοδορίας σας για ένα δευτερόλεπτο. Έγινε η συζήτηση για τον εορτασμό της 20ης επαιτίου του ευρώ, που ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Πάντως, οι έξι ομιλητές που μίλησαν για το, τις επιτυχίες του ευρώ ήταν άνδρες μόνο. Ελπίζω να μην χρειαστεί να περιμένουμε άλλα 20 χρόνια μέχρι ότου συμπεριλάβουμε και τι γυναίκε στη συζήτηση αυτή όπως αξίζει. Ευχαριστώ και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να περάσουμε στι ψηφοφορίε και πριν περάσουμε στι ψηφοφορίε, να κάνω μια ανακοίνωση. Πολλέ επιτροπέ αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικέ διαπραγματεύσει με βάση το άρθρο 69 γ, παράγραφο 1 του εσωτερικού κανονισμού εκθέσει που αποτελούν τις εντολές για τις διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται στην ιστοσελίδα του, της Ολομέλειας και οι τίτλοι τους θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης. Με βάση το άρθρο 69 γ, παράγραφος 2 μέλη ή πολιτικές ομάδες ε, που συγκεντρώνουν το απαραίτητο ελάχιστο κατόφλι μπορούν να ζητήσουν γραπτός μέχρι αύριο, δηλαδή ημέρα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου μέχρι τα μεσάνυχτα, η απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων να τεθεί σε ψηφοφορία. Αν δεν υποβληθεί αυτή η αίτηση για ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, για να τεθεί η απόφαση αυτή σε ψηφοφορία εντό τη προθεσμίας που σα ανέφερα, οι επιτροπέ θα δίνονται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει. Και περνούμε στην ψηφοφορία της έκθεσης ε, Ποσπίσιλ και τον, ε, την ενιαία ε, ψηφοφορία ψηφοφορία μόνο για την έκθεση Ποσπίσιλ θέσπιση στο πλαίσιο του για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται ο κύριος Ποσπίσιλ έχει το λόγο Συγγνώμη, αποσιάζει ο κύριο Ποσπίσιλ, αλλά ζήτησε να αναπευθεί το θέμα στην Επιτροπή. Καλώ, ε, θα το ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε αυτό το αίτημα του κύριου Ποσπισίλ. Διανατάσσεω τη χειρό, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Οπότε, όντω, αναπέμπεται το θέμα στην αρμόδια επιτροπή. Παίρνουμε στην ε, έκθεση Βαλέρο, σύναψη τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αλβανία περί με αντικείμενο δράση που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή στην Αλβανία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση του Κρίστιαν Ταμπρέντα. Πρωτόκολλο Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Κυργιστάν. Προσχώρηση τη Κροατία. Ο κύριος Πρέντα, ο εισηγητής, ε, ζήτησε το λόγο. Όχι, οπότε ψηφίζουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση Πρέντα. Συνολική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυργιζίας. Δεν έχουν υποβληθεί γραπτές αστάσεις βάσει το άρθρο 113 παράγραφος 6, οπότε η σύσταση εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Wim van den Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές. Ενιαία ονομαστική ψηφοφορία. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Monteiro de Aguiar χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές, εμπορευματικέ εμπορευματικές μεταφορές. Τροπολογίες 32 και 33 με ονομαστική κλίση, Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτονται. Τροπολογίες 28 και 34 με ονομαστική κλίση, Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται, εγκρίνονται. Τροπολογίες 29 και 35 και πάλι με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτονται. 30 και 36 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτονται 31 και 37 τώρα με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία τέλος απορρίπτονται και αυτές ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται. Οπότε ολοκληρώσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρώτη ανάγνωση. Περνάμε στην έκθεση Φιέλνερ. Προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένων τρίτων χωρών. Προσωρινή συμφωνία, τροπο, τροπολογία 40, ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41, Διανατάσσεως τη χειρός άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώνει την πρώτη ανάγνωση. Περνάμε στην έκθεση Γκραπίνη, θέσπιση του προγράμματος Τελωνία για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνίων. Ψηφίζουμε την τροπολογία, τις τροπολογίες 1 με 61 μαζί. Διανατάσσει τη χειρό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και ονομαστικά ψηφίζουμε την πρόταση Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Η κυρία Γραπίνη ζήτησε το λόγο. Γραπίνη. Ένα λεπτό ψάχνει ένα μικρόφωνο που να λειτουργεί, κυρία Γραπίνη. μερικές φορές η τεχνολογία μας ξεπερνά. Yeah, we now have a Έχετε μικρόφωνο, τώρα σας ακούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βάσει του ιστορικού κανονισμού ζητώ να αναπευθεί το θέμα στην Επιτροπή για να ξεκινήσουν οι διοργανικές συνεργασίες συζητήσεις. Υπέρ παρακαλώ, για να τα κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση. Πάμε στην έκθεση Χίρμνερ, τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αναπέμπεται, όπως είπαμε στην Επιτροπή. Ξανά, έκθεση Χίρμνερ, τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ονομαστική ψηφορία που ξεκινάει. Πέρας. εγκρίνεται. Πάμε στην έκθεση Μίλνερ ενσωμάτωση διάσταση του φίλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ψηφίσουμε την παράγραφο 6 του αρχικού κειμένου, δυνατά σας τη χειρός, για υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, για ψηφοφορία ψηφοφορίας που ξεκινά, πέρας. εγκρίνεται. Παράγραφος 13 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα, δυνατά στους και τα δύο. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε αν επιτρέπεται, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17 σε δύο τμήματα. Ανατάσσεως χειρός. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ανάταση ισχυρό, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος ξανά άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 21 του αρχικού κειμένου υπέρ παρακαλώ κατά αποχές λυπούμε αλλά πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο ξεκινάει ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Θα το εκτιμούσα αν μπορείτε να σηκώνετε τα χέρια σας. Παράγραφος 24 σε δύο τμήματα. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ανατάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Η ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ανατάσσεως ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 27 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Θα ελέγξουμε την προηγούμενη. Έστω. Έλεγχος για το τρίτο τμήμα της παραγράφου 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ συνάδελφοι, σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Δεν θα κρατήσει πολύ ψηφοφορία. Παράγραφος 27, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28 σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, Νομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα διανομαστικής κλίσεως άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία, την παράγραφο 34, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία, παράγραφος 35, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία, παράγραφος 36, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 39, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Παράγραφο 41 σε δύο τμήματα ανατάσσεως της χειρός. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απόχέ, έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται Παράγραφο 45 του κειμένου υπέρ. Κατά αποχές μικρή διαφορά θα γίνει έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 50 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Μικρότερη διαφορά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μικρότερη, Μικρότερη, μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι πίστευα μάλλον. Παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας. Ψηφίζουμε την τελική σκέψη J, τροπολογία 2, διανατάσεις χειρό χειρός υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ετεολογική σκέψη S, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη U, ανατάσσεται ισχυρό υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη V σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα σύνολό του διανομαστική ψηφορία που ξεκινάει. Πέρασε. και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Πάμε στην έκθεση Μαρινέσκου Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ΆΙΤΕΡ και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύνδεξης. Μία ψηφοφορία έχουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Ψηφίζουμε την έκθεση Hayes, αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Ψηφίζουμε μονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Πάμε στην έκθεση ΞΙΠ, κατευθείαν γραμμή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εντολή του Ειδικού Πεσταλμένου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόθεση τη ελευθερία και τη ελευθερία των πεπιθήσεων εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ματίας και Ουρτασάν ισότητα των φίλων και φορολογικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο παράγραφος 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, να τα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 3 του αρχικού κειμένου θέλετε έλεγχο θα ελέγξουμε λοιπόν την παράγραφο 1 δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται παράγραφος 3 του αρχικού κειμένου διαθέσεις ισχυρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με 4 ψήφους διαφορά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο ε, για την ε, φορολόγηση των επιχειρήσεων ε, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται παράγραφος 13 του αρχικού κειμένου. Εντάξει, έλεγχος για το αρχικό κείμενο, τον υπότιτλο για την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά παρακαλώ βοηθήστε με, σηκώνετε τα χέρια σα. Το αρχικό κείμενο για την παράγραφο 13 ανατάσσεται χειρό υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 14. Ήταν ξεκάθαρο. Τελείωσε ξεκάθαρο. Παράγραφος 14 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17 το αρχικού κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπότιτλος φορολόγηση του κεφαλαίου και του πλούτου υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ονομαστική ψηφοφορία τροπολογία 4 ξεκινάμε πέρας εγκρίνεται Τροπολογία 5, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Παράγραφος 26 του αρχικού κειμένου, διαντάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28 του αρχικού κειμένου, διαντάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, θα γίνει έλεγχος. Άρχεται η ονομαστική κρίση. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 32 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 36 διαντάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7, δυνατά σειρός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφο 41, τροπολογία 8, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Διαντάσει χειρό υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη J, το έχει κειμένο σε δύο τμήματα, δεν ισχυρό, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ, πιο μικρή διαφορά, να κάνουμε έναν έλεγχο, άρχεται η κλίση. Πέρα. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη K, τροπολογία 1